Uh, okay, we, go, ladies and gentlemen. Uh, we have a very... Έχουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, τέσσερα σημεία, δύο ώρες το πρώτο σημείο. Δεν πρέπει να καθυστερήσουμε πολύ. Έχουμε λοιπόν καταρχάς την ανταλλαγή απόψεων για την Προεδρία του G20, την οποία έχει Αργεντινή μαζί με την ΑΦΕΤ αυτό το σημείο υπάρχει μία αντιπροσωπεία στο Κοινοβουλευτικό Φόρουμ στο ε, Buenos Aires από τις 30 Οκτωβρίου μέχρι 2 Νοεμβρίου που θα στείλουμε οι δύο επιτροπές ΑΦΕΤ και ΙΝΤΑ από κοινού. Κύριε Μαρσέλο Σίμα, κάπως έτσι και λυπούμε αν δεν σας πρόφερα σωστά το όνομα. Θα θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε τις προτεραιότητες της ε, Προεδρίας Αργεντινής και ο κ. Αντών Κασάλ από την Προεδρία του Συμβουλίου και από την ΑΦΕΤ έχουμε μαζί μας ε, τον κύριο Κόσο Περμούη, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών, ο οποίος θα είναι ο πρώτος που θα λάβει το λόγο. Έχετε λοιπόν πράγματι το λόγο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω ισπανικά. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Πιντα και ιδίω τον Πρόεδρό τη ε, που κάλεσε στην ανταλλαγή αυτή απόψεων την Επιτροπή Εξωτερικών Είναι πολύ σημαντικό νομίζω να εργαστούμε μαζί στα θέματα αυτά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Είναι θέματα τα οποία υπερβαίνουν το πεδίο αρμοδιοτήτων των ε, μεμονωμένων επιτροπών. Η Αργεντινή ανέλαβε την προεδρία του G20, που είναι το βασικό φόρουμ οικονομική, ε, χρηματοπιστωτική και πολιτική συνεργασία σε διεθνέ επίπεδο για το 2018 και όσο θα έχει την ε, προεδρία η Αργεντινή έχει προγραμματίσει 50 συναντήσεις, μεταξύ των οποίων αυτή των τελών Οκτωβρίου στο Buenos Aires. Σε αυτές τις συνεδριάσεις θα περιλαμβάνονται πολύ σημαντικά θέματα όπως ε, οικονομικά, χρηματοπιστωτικά θέματα που αφορούν την απασχόληση στην ενέργεια ή τη γεωργία. Πολύ ενδιαφέροντα θέματα όλα για τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το όραμα της Αργεντινικής Προεδρίας είναι ε, δημιουργία συνένεσης για μια βιώσιμη δίκαιη ανάπτυξη όπως είχαν ξεκινήσει με το Αμβούργο ε, στη περσινή χρονιά τον Δεκέμβριο που οι ηγέτες αποφάσισαν τη μεγαλύτερη αλληλεγγύη, δικαιοσύνη ε, και ισότητα στον αγώνα για την οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων απασχόληση. Ε, στην ίδια γραμμή, λοιπόν, η Αργεντινή αναζητεί ένα μηχανισμό αναζήτηση συνένεση και έχει εστιάσει τι προσπάθειέ τη στη συγκεκριμένη ε, αναζήτηση ε, τρόπων να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι σε μια σειρά χωρών. Ο πρόεδρος Μαρίθιο Μάκ το Δεκέμβριο του 2017 είχε ζητήσει να υπάρξει διεθνή συνεργασία σε όλες τις πολιτικές, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Η Αργεντινική Προεδρία βασίζεται και στην, και στην βιωσιμότητα που είναι πολύ σημαντικές και ήδη για την εφαρμογή και το σχεδιασμό πρώτα βέβαια των παγκόσμιων κανόνων, που είναι πάρα πολύ απαραίτητοι. Βέβαια ξέρουμε ότι κάποιοι σε αυτόν τον κόσμο δεν θέλουν τους παγκόσμιους κανόνες έτσι, στόχος είναι η αναζήτηση αποτελεσμάτων. Δίκαια και ε, βιώσιμα αποτελέσματα. Στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας, ε, οι πολυμερείς σχέσεις ε, και η παγκόσμια διακυβέρνηση είναι σημαντικό, σημαντικά θέματα εδώ. Έτσι εξηγείται και η παρουσία της Δικής Επιτροπής. Θα συμμετάσχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο Πενοσάρι, στο Κοινοβουλευτικό Φόρουμ στα τέλη Οκτωβρίου και εδώ ολοκληρώνω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος και τώρα το λόγο έχει γι' αυτό εξοχώ της πρέσβης της Αργεντινής. Αν έχετε την καλοσύνη εντός λεπτού και λιγότερο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Σήμα με λένε. Είμαστε Ιταλοί με ισπανική προφορά η απόφαση ή να τα πω ισπανικά. Ε, η απόφαση να γίνει διοργανωθεί η G20 στην, στην Πονος Άιρες ελήφθη στα πλαίσια ε, μιας απόφασης ε, του Προέδρου ε, να ασκήσει εξωτερική πολιτική συμμετοχική και δυνατή. Το G20 έρχεται μετά από τρεις συνεδριάσεις που έγιναν το 2017 στο Buenos Aires. Μία για τις τηλεπικοινωνίες, μία της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας για την Παιδική Εργασία, καθώς επίσης και του ΠΟΕ πάλι σε επίπεδο υπουργικό. Η Αργεντινή έχει και την, πλέον την ε, προεδρία του G20. Όπως πολύ σωστά είπε ο Χαβιέρ, στόχος του G20 είναι να δημιουργήσει συνενέσεις ε, για μια βιώσιμη και δίκαιη ε, ανάπτυξη. Το, η πρώτη σημαντική λέξη είναι η ανάπτυξη, η δεύτερη είναι η ισότητα και η τρίτη είναι η βιωσιμότητα. G20. Ο G20 είναι ο ο οργανισμός που ε, αφορά την ε, οικονομική διακυβέρνηση. Δεύτερο ε, είναι η πολυμέρεια των σχέσεων της Αργεντινής και ο τρίτος λόγος είναι η διάσταση του Νότου. Όπως είπα και προηγουμένως, σε σημαντικό ρόλο παίζει η ανάπτυξη με αυτή η λέξη κλειδί. Νομίζω ότι στη γραμμή και αυτών που είπε ο Χαβιέρα, ε, το σημαντικό είναι να ξέρουμε γιατί μιλάμε, περί ποιου συζητούμε, γιατί συζητούμε γι' αυτά και πώς θα προχωρήσουμε. Building consensus for A fair and sustainable development. Αυτή είναι, ε, αυτός είναι ο τίτλος. Πώς θα το κάνουμε όμως, πώς θα γίνει αυτό στην Αργεντινή. Μέσω τριών προτεραιοτήτων. Το μέλλον της εργασίας. Γνωρίζουμε ότι η τεχνολογική επανάσταση και η παγκοσμιοποίηση αλλάζουν τη μορφή της εργασίας. Ε, κατά την έννοια αυτή η Αργεντινή σε όλη τη διάρκεια του έτους και εξακολουθεί και μέσω του G20 να εργάζεται σε δύο ιδέες. Η νέα παιδεία, η νέα εκπαίδευση, ε, πώς θα προετοιμάσουμε τον κόσμο λοιπόν για αυτό το μέλλον και δεύτερον η τυποποίηση της ε, ε, εργασίας. Πιστεύουμε ότι η τύπη μορφή εργασίας είναι αυτή η οποία δεν οδηγεί στην ε, ε, ανάπτυξη. Επίσης, πάντα για την ε, ανάπτυξη πρέπει να δημιουργηθούν και να οικοδομηθούν αυτές οι υποδομές οι οποίες χρειάζονται έτσι ώστε να κλείσει η ψαλίδα η οποία υφίσταται. Τρίτη προτεραιότητα είναι Sustainable Food for the Future, βιώσιμη, ε, ε, βιώσιμα είδη διατροφής για το μέλλον. Στην ουσία ε, δουλέψαμε για την χρήση της γης και την διατροφική ασφάλεια. Αυτές ήταν ε, οι προτεραιότητες. Όμως, ε, πέρα από αυτές ε, υπάρχουν και άλλα οριζόντια ζητήματα, όπως είναι αυτό του φίλου και διάσταση η οποία θα φαίνεται και στην τελική δήλωση, καθώς επίσης και το θέμα της ισότητας ανδρών και γυναικών, η καταπολέμηση της διαφθοράς και η ενίσχυση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, της συνεργασίας μεταξύ και της σχέσης μεταξύ εμπορίων, εμπορίου και ανάπτυξης. Επίσης, αποφάσεις και ε, ανάληψη ευθύνης όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, θέμα το οποίο βεβαίως ε, ε, ξεπερνά τις χώρες του G20, η Ισπανία, η Χιλή, οι κάτω χώρες η Τζαμάικα, η Ρουάντα και κλπ. είναι χώρες με τις οποίες διευρύνεται αυτή η βάση επί της οποίας στηρίζεται το G20. Πριν ε, ε, τελειώσω την εισαγωγική μου παρουσίαση, θα ήθελα ιδιαίτερος να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ρόλο που ανέπτυξε στην, ε, στον Buenos Aires. Πολλοί επίτροποι της συνεργασίας, της ψηφιακής οικονομίας, της γεωργίας, της βιομηχανίας ταξίδεψαν μέχρι τον Buenos Aires και συνέβαλαν τα μάλα στην επίτευξη συμφωνιών. Θα ήθελα λοιπόν να μεταφέρω την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες της κυβέρνησής μου. Μέσα σε 5 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα ολοκλήρωσα την παρέμβασή μου. Εξαιρετικά λοιπόν, κύριε Πρέσβη. Κύριε Σκασέλα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση κύριε Πρόεδρε. δεν είμαι σίγουρο εάν θα μπορέσω να ξεπεράσω την, τον ενδιαφέρον τη παρουσίαση του κυρίου Πρέσβη, αλλά θα προσπαθήσω. Ακούσατε ποιε είναι οι προτεραιότητε τη ε, Προεδρία του G20 και συμπίπτουν με αυτέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιλαμβάνεστε επίση πόσο σημαντικό είναι αυτή η σημερινή συγκυρία, δεδομένου ότι είναι η δέκατη επέτειο των συναντήσεων των G20 και σε αυτό το πλαίσιο απευθύνουμε μια έκκληση έτσι ώστε να επικρατήσει η πολυμερής προσέγγιση στις διπλωματικές σχέσεις. Όπως έλεγε και ο πρόεδρος Γιούνκερ, αυτό είναι μία από τις βασικές αρχές που θα πρέπει να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε ως Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στη Σύνοδο Κορυφής η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσπαθήσει να ε, υπερασπιστεί το παγκόσμιο, ελεύθερο παγκόσμιο εμπόριο επί τη βάση κανόνων, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα περασπιστούμε λοιπόν την πολυμερή διπλωματία, την διεθνή συνεργασία και για την αντιμετώπιση των παγκοσμίων προκλήσεων. Αυτή είναι η προσέγγιση μας ώψη της Συνόδου Κορυφής. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι την Προεδρία αναλαμβάνει η Αργεντινή, μια χώρα η οποία υφίσταται δυσκολίες από τη σημερινή κατάσταση και έχει την υποστήριξη μας η χώρα στις μεταρρυθμίσεις που προσπαθεί να υλοποιήσει. Ποιε είναι οι προτεραιότητες της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο και είναι προφανές είναι το ζήτημα του εμπορίου. Μετά το, η κλιματική αλλαγή, μετά το μέλλον της εργασίας και η παγκοσμιοποίηση και τέλος η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Πρώτον, όσον αφορά το παγκόσμιο εμπόριο. Το είπα και πριν, ως γενικό στόχο, πιο συγκεκριμένα στην συνάντηση των G20 θα προσπαθήσουμε να υπάρξει αποκλιμάκωση αυτής της σύγκρουσης που διαπιστώσαμε να δημιουργείται τους τελευταίους μήνες, να προχωρήσουμε με θετικές προτάσεις, έχουμε κάνει μια σειρά τέτοιων προτάσεων εμείς, έτσι ώστε να εξυγχρονιστεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και στις τρεις του πτυχές και όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις και όσον αφορά την υποστήριξη και όσον αφορά την επίλυση συγκρούσεων και να βρεθούν ε, λύσεις ε, εν ώψη της Συνόδου στην Οσάκα το 2019 του ΠΟΕ. Πέρα λοιπόν από τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, υποστηρίζουμε τις προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει οι Υπουργοί Εμπορίου για στο πλαίσιο του ΟΣΑ και ελπίζουμε ότι οι ηγέτες της ε, G20 θα ε, δώσουν μια ξεκάθαρη κατεύθυνση για το τι θα πρέπει να γίνει για την, ε, το πλεόνασμα, υπερβολικό πλεόνασμα παραγωγή στο, χάλιβα. Μετά, ήταν πολύ σημαντική αυτή η εβδομάδα η δημοσιοποίηση της, ομάδας ομάδα των Επιστημόνων για το κλίμα από τον ΟΗΕ, Λίγε ημέρε πριν τη συνάντηση του Κατόβιτσε. Και Γνωρίζουμε όλοι ποιε είναι οι επιπτώσει τη κλιματική αλλαγή ε, για την οικονομία μα, για του πολίτε μα. Επομένω, θα συνεχίσουμε να τονίζουμε πόσο σημαντικό είναι να εφαρμοστεί στην πράξη η Συμφωνία των Παρισίων, καθώ επίση και οι στόχοι τη χιλιετία και η Ατζέντα 2030, καθώ επίση και η εταιρική σχέση για την Αφρική. Επόμενο θέμα είναι το μέλλον της εργασίας και η αντιμετώπιση της παγκοσμιοποίησης. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πολλές φορές αναφερθεί στην καλή χρήση, την αξιοποίηση των θετικών της παγκοσμιοποίησης που επηρεάζει πολλές τομείς της οικονομίας. Αυτό σημαίνει ενίσχυση της ισότητας, ε, να επενδύσουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και για καθένα, καθεμιά από τις κυβερνήσεις που εκπροσωπούνται στην G20 αυτό σημαίνει συγκεκριμένους ε, στόχους που θα συζητηθούν και αυτοί στη διάσκεψη της ΟΣΑΚΑ. Θα αναφερθούμε επίσης και στο ζήτημα της φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας. Αυτό είναι ένα τομέα στον οποίο έχουμε πρωταστατήσει ως Ευρωπαϊκή Ένωση με σχετικές ρυθμίσεις και προσπαθούμε να προωθήσουμε και αντίστοιχες διεθνείς πρωτοβουλίες. Μετά θα ζητήσουμε την πλήρη υλοποίηση της που έγινε πέρυσι για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η οποία συνοδεύεται από μια προσέγγιση με τρεις πυλώνες ανάμεσα στους οποίους είναι η καταπολέμηση της ρουζουρπαστικοποίησης και της ρητορικής του μίσου στο ίντερνετ και η διεθνή συνεργασία. Ε, θα προσπαθήσουμε να, να προχωρήσουμε περισσότερο και σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Το συγγνώμη που ξεπέρασα λίγο το χρονικό μου όριο. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφοί μου τώρα έχουν το λόγο αν κάποιος θέλει. Ο κύριος Βίνκλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την αυτοξόφατα τον Πρέσβη για την παρουσία των στόχων. Ε, ε, Είπατε κάτι και με αυτό θα ε, ξεκινήσω. Μιλήσατε για δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό είναι το μότο τη Αργεντίνικη Προεδρία. Ακριβώ αυτό μα ενδιαφέρει στην Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου. Και ο στόχο είναι να υπάρχει συνεργασία ε, στα εμπορικά ζητήματα και στα ζητήματα των επενδύσεων. Συνεργασία λοιπόν είναι η λέξη κλειδί και ξέρουμε ότι είναι μοχλό ανάπτυξη ε, το εμπόριο. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε βιώσιμο εμπόριο, πρέπει να λειτουργεί σωστά το διεθνέ καθεστώ εμπορικών συναλλαγών και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε μια στο δυνατόν πιο ισορροπημένη κατανομή του κόστους αλλά και των ωφελιών του εμπορίου αυτού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το είπε και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, έχει συνεπείς και συνεκτικές προτάσεις πριν από λίγες εβδομάδες στη Γενέβη, τέλη Σεπτεμβρίου. Δημοσιοποιήθηκαν, έχουμε ένα πακέτο λοιπόν προτάσεων και ελπίζουμε να έχει απήχηση και να βρει και στήριξη μεταξύ των άλλων μελών ε, και στην ομάδα του Τζέιτ 8 και Ξέρουμε ότι υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην παγκοσμιοποίηση και στο εμπόριο, άρα πρέπει να πανεργοποιήσουμε την όλη συζήτηση για την αποτελεσματικότητα του εμπορίου και το ότι είναι δίκαιες όλες αυτές οι εμπορικές συμφωνίες. Φυσικά επίσης ότι πρέπει να προωθήσουμε περισσότερο επενδύσεις και εμπορικούς δεσμούς. Ο προστατευτισμός δεν έσωσε ποτέ κανέναν. Ούτε έλυσε και κανένα πρόβλημα στον κόσμο. Επομένω, οι εμπορικοί πόλεμοι δεν έχουν νικητέ. Κάποιε πρωτεύουσε από την άλλη πλευρά του ανού μπορεί να έχουν μια διαφορετική άποψη. Δεν ισχύει όμω αυτό και πρέπει να πω ότι και στο πλαίσιο τη ομάδα των 20 θα πρέπει να προωθήσουμε τι ιδέε αυτέ και να ε, ζητήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερε πολυμερει φορέ να απογράφονται ή αλλιώ ε, διμερεί, που να είναι όμω συμπληρωματικέ προ τη φύση του. Το μήνυμά μας λοιπόν ω αντιπροσωπεία που θα συμμετάσχει σε αυτό το κοινοβουλευτικό φόρουμ ε, στη, στο Buenos Aires ε, είναι ότι μόνο με τη συνεργασία μπορούμε να δημιουργήσουμε βιώσιμη, ισορροπημένη ε, για όλους ανάπτυξη που θα δημιουργεί θέσεις εργασίας και θα ευνοεί τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, Κάποιος άλλος? Κάποιος συνάδελφος από τους βουλευτές, ο κύριος Darthmouth. Ευχαριστώ. Θα με ενδιαφέρει να ακούσω την άποψη του προεδρεύοντος ε, της G20 για τη Ρωσία και τις, ε, και τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία και θα ήθελα να μας πει επίσης την άποψή του για το Ιράν και τις κυρώσεις κατά του Ιράν. Πολύ σύντομο το σχόλιο Άρα δύσκολα θα το παρακάμψει ο Προεδρεύων. Ελπίζω να μου δώσει σαφείς απαντήσεις. Άλλος κανείς, λέει ο Πρόεδρος. Όχι, δεν βλέπω κάποιον άλλον θέλει το λόγο. Κύριε Πρέσβη, θα θέλετε να απαντήσετε σε αυτή την πολύ σύντομη ανταλλαγή απόψεων. Και με ο κύριο Κασέλ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ εύκολο να απαντήσω στον ε, συνάδελφοι που είναι στο βήμα, που είναι στο Προεδρείο, ε, γιατί δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω απόλυτα. Το προσπαθήσαμε και τον δοκιμάσαμε τον προστατευτισμό για δεκαετίες στην Αργεντινή. Δεν λειτουργήσε, άρα εμπειρία έχουμε. Εγώ ήμουν στη Γενέβη ως πρέσβης και εκεί πιέσαμε ε, το πολυμερές θεματολόγιο να υποστηριχθεί. Το ίδιο θα κάνουμε στην Αργεντινή. Μην ανησυχείτε καθόλου γι' αυτό λοιπόν γιατί πιστεύουμε πραγματικά ότι αυτός είναι ο δρόμος προς τα εμπρός, διότι πιστεύουμε ότι το εμπόριο δημιουργεί πλούτο. Οι προηγούμενε κυβερνήσει στην Αργεντινή μάλλον δεν πίστευαν το ίδιο, αλλά εμεί αυτό πιστεύουμε. Σε ό,τι αφορά το άλλο ερώτημα, όμω δεν μπορώ να το απαντήσω. Ευχαριστώ. Thank you. And, uh, then the commission, if, uh, Ευχαριστώ. Η Κομισιόν, κύριε Κασέλ, θα θέλατε κάτι να πείτε. Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε. Γιατί φυσικά και είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο με τον προλαλήσαντα. Και συμφωνώ, σας ανέφερε και στις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε και δεν μπορώ να επαναλάβω τη σημασία που έχει συλλογικότητα η συνεργασία. Γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Άρα δεν έχω να πω τίποτα διαφορετικό. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Άρα ολοκληρώνεται το σημείο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την αφήξω τον πρέσβη για την παρουσία του εδώ. Και βέβαια, εμείς θα πάμε στον Πενοσάιρες και θα συμμετάσχουμε σε αυτό το κοινοβουλευτικό φόρουμ της ομάδας των 20. Το περιμένουμε πώς και πώς. Προχωράμε γιατί είμαστε υπό μεγάλη πίεση χρόνου. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε ευθύ αμέσω στο σημείο 11 τη μερσιά διάταξη, που είναι ανταλλαγή απόψεων για τι εμπορικέ σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία τη Νοτιοαφρική. Να καλωσορίσω ε, τους εκπροσώπους ε, του, τα της πρεσβείας, την προσωπή λοιπόν από την πρεσβεία της ε, Νοτιοαφρικής Ο πρέσβης νομίζω, ο ίδιος... Ε, Again, I apologize. Σανκού είναι εδώ. If not, then uh, you can correct me later. Ελπίζω να το πρόφερα σωστά, αλλιώ διορθώστε με. Η πταμελής αντιπροσωπεία της ΙΝΤΑ θα μεταβεί στην Νότια Αφρική στα τέλη Οκτωβρίου για να δει πώς προχωρά η υλοποίηση της ε, οικονομικής εταιρικής σχέσης. Δύο χρόνια πάνε από τότε που τέθηκε σε Θα συζητήσουμε επίσης ε, με τους ομολόγους μας και τα ε, μερή ζητήματα. και τις εμπορικές μας σχέσεις. Πέρασε καιρός που είχαμε συζήτηση για τα θέματα των εμπορικών